Θα ξεκινήσουμε εκ νέου τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδριάσεως και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στα πρακτικά είναι διαθέσιμα. Δεν έλαβα υπόψη κανένα σχόλιο. Ούτε βλέπω κάποιον που θέλει να μιλήσει για το θέμα αυτό. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι εγκρίθηκαν. Θα μπούμε